One minute. Άρχεται η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτική Ανάπτυξης. Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω όλους θερμά και ιδιαιτέρως να καλωσορίσω τον κύριο Χόγκαν σας καλωσορίζω κύριε Χόγκαν εκ μέρους όλων των μελών της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης. Η παρουσία σας ε, αναφυσβήτητα αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην Επιτροπή μας και ευελπιστώ ότι θα αποτελέσει και την απαρχή μιας καρποφόρας συνεργασίας που θα συμβάλλει στην προάσπιση και την ανάπτυξη μιας ισχυρής ε, και βιώσιμης ε, καθώς και ισορροπημένης ευρωπαϊκής γεωργίας. Θα ήθελα λοιπόν να καλωσορίσω όλους τους παρόντες, ε, τους καλεσμένους μας, τους εκπροσώπους της Γενικής Επιτροπής, τους υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης και φυσικά τα μέλη της Επιτροπής μας. Να πω δύο λόγια για τον υποψήφιο επίτροπό μας. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Κόρκ, ανέλαβε την οικογενειακή εχρωτική εκμετάλλευση ο κύριος Χόγκαν και κατόπιν ίδρυσε το δικό του ε, ε, μεσητικό και ασφαλιστικό γραφείο. Από το 1983 εξελέγει στο Δημοτικό Συμβούλιο του Κιλκένη για πρώτη φορά. Έκτοτε συγκέντρωσε πλούσια πολιτική πείρα. Στην αρχή δραστηριοποιήθηκε σε τοπικό επίπεδο και κατόπιν εξελέγει γεροσιαστής και βουλευτής από το 1987 και έκτοτε. Διατέλεσε και υπουργό Περιβάλλοντος, Κοινοτήτων και τοπικής, τοπικών αρχών και τοπικής διακυβέρνησης από το 1211 έως το 1214. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με βάση τις κατευθυντήριες γραμμές για την έγκριση της ε, Επιτροπής που περιλαμβάνονται στο παράρτημα 16 του εσωτερικού μας κανονισμού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει τους υποψηφίους επιτρόπους με βάση τη γενική τους ε, ε, επάρκεια, την προσήλωσή τους στην ευρωπαϊκή ιδέα και την προσωπική τους ανεξαρτησία. Επίσης θα αξιολογήσουμε και τις γνώσεις τους σε σχέση με το χαρτοφυλάκιό τους καθώς και τα επικοινωνιακά τους προσόντα. Θα ήθελα επίσης να σας υπενθυμίσω ότι πριν την ακρόαση ο προτινόμενος επίτροπος Φιλ Χόγκαν απέστειλε γραπτός απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο. Οι γραπτές αυτές απαντήσεις σας έχουν μοιραστεί και μάλιστα μεταφρασμένες σε όλες τις επίσημες γλώσσες σε ό,τι αφορά τη διάρθρωση της συζήτησης. Θα ήθελα να σας επισημάνω μερικά σημαντικά διαδικαστικά σημεία. Ο υποψήφιος ε, Επίτροπος θα λάβει το λόγο για μια εισαγωγική παρουσίαση που δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Στο τέλος της συνεδρίασης θα έχει άλλα 5 λεπτά για τελικά σχόλια. Μετά την εισαγωγική αυτή παρουσίαση θα έχουμε χρόνο για να υποβάλουμε 45 ερωτήσεις θα γίνει συζήτηση με βάση την αρχή του ping-pong. Δηλαδή, θα υποβάλλετε μία ερώτηση μονόλεπτη και θα δίνετε μία δίλεπτη απάντηση. Ένα τρίλεπτο λοιπόν για κάθε έρωτα απάντηση. Επειδή το θέμα είναι πολύ σημαντικό, θα είμαι πολύ αυστηρό στην τήρηση του χρόνου. Είναι σημαντικό αυτό για την εύρυθμη διεξαγωγή της ακρόασης. Θα σας θερμοπαρακαλούσα λοιπόν να τηρήσετε όλοι ευλαβικά το χρόνο σας, το χρόνο μιλίας που έχει ο καθένας. Προβλέπετε μία ανοχή 5 δευτερολέπτων για υπέρβαση του χρόνου μιλίας από τους ευρωβουλευτές και 10 δευτερολέπτων ανοχή για υπέρβαση του χρόνου μιλίας από τον υποψήφιο επίτροπο. Μετά την παρέλευση αυτών των 5 και 10 δευτερολέπτων θα απενεργοποιώ το μικρόφωνο. Μάλιστα θα ανάψει ένα φως ε, μπροστά σας 10 ε, δευτερόλεπτα πριν την πάροδο του χρόνου που δικαιούστε. Είναι σημαντικό να σεβαστούμε όλους αυτούς τους κανόνες ε, προκειμένου να προλάβουν όλοι οι ευρωβουλευτές να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους στον προτινόμενο επίτροπο. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι προβλέπεται διερμηνία σε 24 γλώσσες και τα Ιρλανδικά. Όλοι μπορούν να μιλάνε και να ακούν τη γλώσσα τους. Αλλά σας υπενθυμίζω ότι επειδή υπάρχει διερμηνία, καλό θα ήταν να, ε, να μην μιλάτε πολύ γρήγορα. Επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η ακρόασή μας μεταδίδεται ζωντανά μέσω διαδικτύου στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στον ίδιο ιστότοπο θα βρείτε αργότερα και την ε, μαγνητοσκοπημένη αναμετάδοση της ακρόασης. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο κυρίως θέμα. Και με βάση το πρόγραμμα και το χρονοδιάγραμμα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον προτινόμενο μας επίτροπο, τον κύριο Χόγκαν, και να του δώσω το λόγο για την εισαγωγική του παρουσίαση που, όπως τον παρακάλεσα και στην αρχή, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το τέταρτο.